5 25 Μαρτίου 2010, 9 με 1 το πρωί. Έχει δημοσιευτεί η ημερησία διάταξη. Μπορεί να τη διαβάσετε στη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να σε όλους τους συναδέλφους, ε, να τους ευχαριστήσω που ήταν εδώ και επίσης τους διερμηνείς που άντεξαν. Ευχαριστώ.